εύχομαι επί της διαδικασίας πάλι. Ελπίζω να είναι επί της διαδικασίας. Ευχαριστώ πρόεδρε θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους. Να πω επίσης ότι παραδοσιακά οι συζητήσει για τα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητιούνται Παρασκευή απόγευμα, μα είναι πάρα πολύ σημαντικές όμες και θα έπρεπε να ψηφίζονται από μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών. Ελπίζουμε στην επόμενη θητεία να αλλάξει η παράδοση αυτή να συζητούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα το πρωί ούτω ώστε να μην είναι μονάχα 30 βουλευτές παρόντες όταν κουβεντιάζουμε τόσο σοβαρά θέματα ναι βεβαίως κατάλαβα τι μας είπατε και το σημειώσαμε αλλά Βεβαίω, επειδή είναι πέμπτη απόγευμα, δεν σημαίνει ότι αυτοί που ενδιαφέρονται δεν μπορούν να έρθουν. Δεν μπλοκάρουμε, δεν εμπιδίζουμε κανένα να έρθει. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας, πέρα στη συνεδρίαση.